ομιλιών ενό λεπτού βάσει του άρθρου 163. Η επόμενη συνεδρίασή μα λαμβάνει χώρα αύριο από τι 9 ω τι 2 και από τι 3 ω τι 8.30. Η ημερήσια διάταξη βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού.